και ελπίζω ότι θα μπορέσω να κάνω και εγώ ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Άστον, κλείνει η συζήτηση αυτή. Περνάμε τώρα στην δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπα του εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, για τη ε, θέση σε ισχύ της σύμβασης. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σα είμαι ιδιαίτερως ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να συστήσω το θέμα αυτό για τα όπλα διασποράς. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό, σημαντική στιγμή ε, μερικούς μήνες πριν από θέση ισχύ τη σύμβαση για τα όπλα διασποράς. Ε, η σύμβαση αυτή θα προλάβει τη χρήση, την αποθήκευση και την παραγωγή των όπλων διασποράς. Όπως έγινε με, τα, με τις νάρκες κατά προσωπικού, η, τα όπλα διασποράς εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους για, την, για τους πολίτες και επηρεάζουν ιδιαίτερα τα παιδιά. Η φύση ακριβώς των όπλων αυτών ε, βαίνει κατά των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών όχι μόνο εκλείουν ε, εκρηκτικά υλικά βόμβες ε, σε ε, ευρύτατες περιοχές χωρίς διακρίσεις αλλά μπορούν να κραγούν ανα πάσα στιγμή ακόμα και δεκαετίες μετά το πέρας μιας σύραξης. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να πετύχει μια πλήρη απαγόρευση αυτών των θανατηφόρων όπλων. Η Σύμβαση για τα όπλα διασπορά συμφωνήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 και μόνο σε 1,5 χρόνο 106 χώρες την υπέγραψαν και 36 την επικύρωσαν. Η... Ε, αναμένουμε μια σημαντική πρόοδο να γίνει στις κοινέ μας προσπάθειες να μειωθούν να μειωθεί και να απαγορευτεί η παραγωγή, η χρήση και η μεταφορά των πυρομαχικών διασπορά. Αξιότιμα μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη δεσμεύεται απολύτω στο να αντιμετωπίσει τι επιπτώσει των όπλων διασπορά στου πολίτε μέσω όλων των ε, μέσων των εργαλείων που έχει στη διάθεσή τη. Παρόλο που δεν είναι όλε οι χώρε μέλη τη σύμβαση. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δραματίσει ένα ρόλο σε αυτό το πεδίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υποστηρίζει τις ευρύτερες, τη διεύρυνση των διαπραγματεύσεων για ένα επιπρόσθετο πρωτόκολλο για τα όπλα διασφοράς στη Σύμβαση των Ηνωμένων Αθηνών για τη χρήση ορισμένων σημαντικών όπλων. Ο στόχος εδώ είναι να διευρυνθεί ε, το όργανο αυτό και να περιληφθούν ακόμα περισσότερες χώρες. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πολύ ξεκάθαροι προς το σημείο αυτό. Η σύμβαση για τη χρήση ορισμένων συμβατικών όπλων είναι μια σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και γι' αυτό είναι πραγματικά πολυμερές εργαλείο ε, το οποίο γίνεται μου διαπραγμάτευση σε ένα ευρύτερο φόρουμ. Οι διατάξει και αυτέ του επιπρόσθετου πρωτοκόλου συμβάλλουν στη μείωση των ε, ε, επιπτώσεων για τον άμαχο πληθυσμό. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοστεί αυτό το πρωτόκολλο και το η σύμβαση για το πρόσθετο πρωτόκολλο. Και αυτό ακριβώς κάνουμε μια κοινή δράση που στηρίζει την καθολικοποίηση τη σύμβαση και την πλήρη τη εφαρμογή. Στι διαπραγματεύσει για το πρόσφατο πρωτόκολλο για τα πυρομαχικά διασπορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί την απαγόρευση, όχι μόνο τη μείωση, τη χρήση τη παραγωγή ε, και τη αποθήκευση ορισμένων πυρομαχικών ε, διασπορά. Εγώ αναγνωρίζω ότι το εύρο αυτού του πρωτοκόλλου δεν μπορεί να είναι τόσο ευρύ όσο η σύμβαση για τα ε, πυρομαχικά διασπορά, αλλά μπορούμε να πετύχουμε ένα ένα πρωτόκολλο, μια ευρύτερη συμμετοχή, ιδιαίτερω εκείνων των χωρών μελών που παράγουν και αποθηκεύουν αυτά τα όπλα. Αυτό θα μα βοηθήσει να προσεγγίσουμε περισσότερο του στόχου μα. Όσον αφορά τα περαιτέρω βήματα για τη σύμβαση για τα όπλα διασπορά, χαίρομαι που έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίε για την πρώτη συνάντηση των συμβαλόμενων μερών που θα λάβει χώρα το 2010. Η συνδιάσκεψη του Σαν Διέγκο τον Ιούνιο έδειξε το υψηλό επίπεδο δέσμευσης πολλών χωρών όπως ε, συνέβη ε, επίσης και για τους, όπως και για τους εκπροσώπους των ε, μη κυβερνητικών οργανισμών. Και θα ήθελα να δώσω τώρα μια έφαση στο γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά ανέλαβε ένα ιδιαίτερο ενεργό ρόλο. Συνδράμουμε τι τρίτε χώρε να απαλλαγούν από τα κατάλοιπα αυτών των όπλων διασπορά να καθαρίσουν τις περιοχές και να παράσχουν συνδρομή στα θύματα στο Αφγανιστάν όπως το Λάο, την Καμπότζη, το Λίβανο ή το Σουδάν. Τα τελευταία δέκα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε, έδωσε 300 εκατομμύρια ευρώ ε, ε, στο, για, το, για, την, ε, για τον καθαρισμό από τις νάρκες κατά προσωπικού. Αξιότιμα μέλη αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη συζήτηση. Ε, ευχαριστώ κυρία Άστον. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκαλέρ για Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ πολύ κυρία είπατε εκπρόσωπα για τα εισαγωγικά σας λόγια. Υποστηρίζω πλήρως τα όσα είπατε και πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε το τι έπραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την απομάκρυνση από αυτά τα όπλα. Η πόλεμοι είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο τόσο για τους εμπλεκόμενους πολίτες, αλλά εντός αυτού του κακού σενάριου υπάρχει ένα είδος ακόμα πιο θανατηφόρων όπλων όπως είναι αυτά τα πυρομαχικά διασποράς που μπορούν να αναπτύξουν τις ολέθριες επιδράσεις τους για πολλά χρόνια. Γι' αυτό είναι σημαντικό από τη μία την 1η Αυγούστου να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ότι η σύμβαση αυτή πράγματι τίθεται σε ισχύ και από την άλλη είναι μια σημαντική ευκαιρία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει ιδιαίτερος ούτε ώστε να φροντίσουμε για την τάξη στο δικό μας σώμα. Δηλαδή συγκεκριμένα να καλέσουμε εκείνες τις χώρες μέλη που μέχρι στιγμής δεν έχουν ε, είτε υπογράψει είτε επικυρώσει ε, τη σύμβαση, να καλέσουμε τις χώρες μέλη να το πράξουν το συντομότερο, λέμε μέχρι τέλος του χρόνου. Υποθέτω ότι μέχρι την 1η Αυγούστου θα ήταν πραγματικά ευκταίο, παρόλο που ίσως δεν είναι εφικτό γιατί κάποια κοινοβούλια έχουν θερινές διακοπές. Ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε επίσης είναι η αυγουστου θα ηταν πραγματικα ευκταιο παρολο που ισως δεν ειναι εφικτο γιατι καποια κοινοβουλια εχουν φερνες διακοπες ενα θεμα το οποιο αναφερθηκε επισης ειναι η έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει ένα νομικό πρόσωπο να προσχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση. Ίσως αυτός είναι ένας ε, τρόπος να ε, ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη να το πράξουν αυτό διμερώς. Εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα και να λάβουν ένα πρωτοπόρο ρόλο έναντι των τρίτων χωρών ούτως ώστε να τις βοηθήσουν να απαλλαγούν από τα κατάλοιπα των όπλων των πυρομαχικών διασποράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Κύριε Γκόμες για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Οι βόμβες διαφοράς δεν κάνουν καμία διάκριση μεταξύ των στόχων. Όλα αυτά αντίκειται στο διεθνές ε, δίκαιο και στην παγκόσμια ασφάλεια. Τα βασικά θύματα αυτών των όπλων διασποράς είναι από όμενες χώρες. Η σύμβαση υποχρεώνει τις χώρες μέλη να καταστρέψουν το πλωστάσιό τους, να καταστρέψουν τα όπλα, τις βόμβες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και να προστατεύσουν τα ε, θύματα. Η σύμβαση τίθεται σε εφαρμογή στην 1η Αυγούστου και μόνο 16 χώρε την έχουν κυρώσει. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειε για να βάλουμε κάποιο τέλο στη μεταφορά αυτών των όπλων. Εννέα χώρε της Ευρωπαϊκή Ένωσης δεν έχουν ακόμα κυρώσει τη σύμβαση η χώρα μου, η Πορτογαλία ήταν ε, μία από εκείνες τις χώρες που υπέγραψαν το Δεκέμβριο του 2008 τη σύμβαση δύο χρόνια. Μετά δεν έχει ακόμα γνωμοδοτήσει το Κοινοβούλιο η τα αυτή μας φέρνει πραγματικά σε δύσκολη θέση. Η γυναία Πισάου δήλωσαν ότι η κύρωση θα γίνει τον επόμενο Αύγουστο, πριν δηλαδή από την Πορτογαλία. Αυτά, αυτό είναι απαράδεκτο, γι' αυτό το λόγο θα παρακαλούσα την ε, κυρία Άστο να προβλέψει μια κύρωση για αυτούς που δεν ε, θα κυρώσουν ε, τη σύμβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο και οι επτά χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση θα πρέπει να αναλάβουν τις ε, ευθύνες τους. La parole est à Madame Lynn pour 3 minutes. Κυρία Λίν, Οι βόμβες διασποράς έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά θύματα και συνεχίζουν να δημιουργούν. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι τα περισσότερα θύματα είναι παιδιά. Ας ε, σκεφτούμε την περίπτωση ενός μικρού κοριτσιού από το Βιετνάμ που έχασε και τα δύο της πόδια. Η τραγωδία είναι ότι το κοριτσάκι αυτό θεωρήθηκε τυχερό. Τα περισσότερα ατυχήματα καταλήγουν σε θανάτους. Μετά από χρόνια εξρατείας τώρα υπάρχει μία σύμβαση που μας επιτρέπει να επιφέρουμε αλλαγέ. Είναι ζωτική σημασία πρωτίστως όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπογράψουν και να κυρώσουν τη σύμβαση κατεπηγόντως όπως είπε η κυρία ε, Μόνο 11 χώρες μέλη κύρωσαν την σύμβαση μέχρι στιγμής. Σε λίγο θα τεθεί ενισχύ η σύμβαση αυτή και θα ήθελα να πω ότι απαιτείται μια συντονισμένη προσπάθεια από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για να πιστούν όλε οι χώρε μέρη για να υπογράψουν και να κυρώσουν. Οι χώρε μέρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που υπέγραψαν θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν για να εφαρμόσουν εθνική νομοθεσία, για να μπορέσουν να καταστρέψουν τα αποθέματα όπω έχει ήδη κάνει η Ισπανία. Το 2002 ήμουν εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για την ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών τα δικαιώματα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίε. Αυτή υιοθετήθηκε το 2006. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα υπογράψει αυτή τη βασική σύμβαση. Θα είναι σαφώ μία αντίφαση αν δεν τα καταφέρουμε να δραστηριοποιηθούμε για τι βόμβε διασπόρά. Είναι σημαντικό, κοιτάζοντα προ το μέλλον και το Συμβούλιο και η Επιτροπή, να συμπεριλάβουν την απαγόρευση των όπλων διασπορά σε μια συμφωνία με τι τρίτε χώρε. Και θα επιθυμούσα να ακούσω τα προγράμματα τη ΥΠΑ εκπροσώπου η σύμβαση αναφέρεται σε ένα νέο ανθρωπιστικό πρότυπο για βοήθεια στα θύματα στο άρθρο 5. Ζητά βέλτικες πρακτικές και ε, κατευθυντηρίους ε, γραμμές, ε, η ψυχολογική υποστήριξη από κατάσταση. Επίσης σημαντικό, όπως είπε η κυρία Άστον, είναι η απαλλαγή από εκατομμύρια βόμβες διασποράς. Το άρθρο 6 τη σύμβαση ζητάει από κάθε χώρα να παράσχει βοήθεια για την καταστροφή των όπλων διασποράς και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα μέσα και τις τεχνολογίες που αφορούν την απαλλαγή από αυτά τα όπλα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σώσουμε τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί. Ξέρουμε τις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα όπλα. Τα γνωρίζουν ε, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση. Σας ζητώ, όλου, ζητώ από όλους σας να υποστηρίξετε αυτή τη ε, σύμβαση. Η κυρία Λούνατσεκ έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Άστον, κυρίες και κύριοι για πρώτη φορά πριν από τέσσερα χρόνια ασχολήθηκα με το θέμα αυτό των όπλων διασποράς όταν μια ομάδα της κοινωνίας των πολιτών ε, απευθύνθηκε στο Αυστριακό Κοινοβούλιο και μας ζήτησαν να κάνουμε μια διοργάνωση για να προετοιμάσουμε τη σύμβαση. Ήταν ε, άνθρωποι που ίδιοι είχαν χάσει ένα πόδι, ήταν ανάπηροι από αυτά τα όπλα, είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας και μας έδειξαν ε, τι συμβαίνει όταν ε, κρύγνεται μια τέτοια βόμβα. Είναι διάφορα χρωματιστά μικρά κομμάτια τα οποία διαχέονται και παραμένουν για χρόνια εκεί. Παιδιά τα οποία αργότερα πάνε να παίξουν εκεί και βλέπουν αυτά τα πολύχρωμα κομματάκια, τα παίρνουν στα χέρια, εκρήγνεται και χάνουν το ένα πόδι χέρι τους. Αυτό με εντυπωσίασε τότε τόσο πολύ που άρχισα να στατεύουμε για την υπόθεση αυτή στην Αυστρία. Ε, ε παρόλο που η χώρα μου τόσο, ήταν μια από τις πρώτες που προσεπέγραψε και κύριο στη σύμβαση. Αλλά πολλές χώρες δεν το έκαναν και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορέσαμε με αυτό το ψήφισμα να κινητοποιήσουμε πέντε πολιτικές ομάδες να το στηρίξουν. Και αυτό θα ήθελα να το πω ειδικά στον κύριο Γκάλερ, όπου η πολιτική του ομάδα είχε πολλές επιφυλάξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καταφέρετε να κινητοποιήσετε και τη δική σας πολιτική ομάδα, να κατονομάσετε εκείνες τις χώρες που ακόμα δεν έχουν προσυπογράψει και κυρώσει τη σύμβαση και που δεν είναι διατεθειμένες πραγματικά να καταστρέψουν τα αποθέματα των όπλων αυτών και που δεν θα το κάνουν ποτέ. Κυρία Άστον, δύο συγκεκριμένα ερωτήματα προς εσάς. Το αίτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφορήσει σε αυτή τη σύμβαση ως ίδιο ε, νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες για να προσθέσει στις διαπραγματεύσεις αυτές ε, ε, τον όρο καταστροφής των καταλήπων των πυρομαχικών διασποράς. Προτίθεστε να το κάνετε. Ευχαριστώ κυρία Λούνα Τσέκ. Η κυρία Λόζινγκ, δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους προλύσαντες ε, και θα ήθελα να τους πω ότι συμφωνώ μαζί τους. Ε, πραγματικά τα, οι βόμβες διασποράς είναι τα πιο, από τα πιο βία όπλα που υπάρχουν. Μέχρι πρόσφατα ε, χρησιμοποιούν τόσο από τι ΗΠΑ όσο και από χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, στη Ιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και στην Ιεμένη. Χρησιμοποιήθηκαν ευρύτερα. Και είναι φρικιαστικό ε, το τι έγινε ε, με τα θύματα. Κατά 98% τα θύματα είναι άμαχος πληθυσμός και από αυτούς 20% είναι παιδιά. Τώρα, πώς ε, χαράσετε η προοπτική της περαιτέρω χρήσης αυτών των όπλων και πώς μπορούμε να την αξιολογήσουμε. Είναι αξιοσημείο το γεγονό ότι η Deutsche Bank μέσω θηγατρικών συμμετέχει ή επενδύει στην παραγωγή αυτών των δολοφονικών όπλων. Οι σχέσεις της Deutsche Bank προς τους ε, προμηθευτές ε, με τη Lockheed για παράδειγμα έχουν αποδειχθεί. Θεωρώ ότι είναι πονίδιστο συνειδητά να θέλει κανείς να κρατήσει χρήματα με το θάνατο των αμάχων. Η χρήση, η παραγωγή, η αποθήκευση και η μεταφορά αυτών των όπλων θα πρέπει να απαγορευτεί και επίσης ε, δεν θα πρέπει να γίνονται συναλλαγές και επιχειρήσεις με αυτά τα όπλα. Όλες οι χώρες μέλη ε, ε, θα πρέπει να υπογράψουν ε, τη σύμβαση αυτή πριν από την 1η Αυγούστου αυτού του έτους. Και εάν αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει την 1η Αυγούστου, το ταχύτερο δυνατό, όπως είπε και ο κ. Γκάλερ. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ένα μορατόριο για τη χρήση, την παραγωγή και την μεταφορά των ε, όπλων ε, διασποράς μέχρι την κύρωση τη σύμβαση. και το ταχύτερο δυνατό θα πρέπει να καταστραφούν τα αποθηκευμένα όπλα. Χαίρομαι πάρα πολύ και θα ήθελα να χαιρετήσω εξ ονόματο της ΓΚΟΕ αυτό το ψήφισμα, αυτή τη συνεργασία που έγινε μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων για την υποστήριξη του κοινού ψηφίσματος για τη σύμβαση αυτή. Και θεωρώ το ψήφισμα αυτό ε, συνιστά μια μεγάλη επιτυχία στον αγώνα κατά αυτού του δολοφονικού όπλου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λόζινγκ. Ο κύριο Σμιθ δεν παρίσταται, άρα θα περάσουμε άμεσα στη δικασία Catch the Eye και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Παπα-Νικολάου για ένα λεπτό. Δεν βρισκόμαστε κατά από ιδιαίτερη πίεση χρόνου, δεν είμαστε ιδιαίτερως πολύ άρα. Πράγματι, υπόθηκε από του συναδέλφου. μόνο 11 κράτη-μέλη στα 27 έχουν κυρώσει αυτή την τόσο σημαντική συνθήκη για την ε, κατάργηση της χρήσης, παραγωγής και αποθήκευση και μεταφοράς όπλων διασποράς και κανείς δεν διαφωνεί ότι πρέπει να επιδιώξουμε όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν αυτή τη συνθήκη. προκύπτει βεβαίως το ερώτημα γιατί τα υπόλοιπα κράτη μέλη δεν έχουν κυρώσει μέχρι σήμερα τη συνθήκη παρότι η έναρξη είναι στην 1η αυγούστου. η κύρια αιτιολόγηση είναι λόγοι εθνική ασφάλεια, και σε μεγάλο βαθμό σε κάποιε περιπτώσει είναι δικαιολογημένη ιδιαίτερα μάλιστα όταν γειτονικά κράτη εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζουν αυξημένη επιθετικότητα κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι αν θέλουμε πραγματικά όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν αυτή τη συνθήκη και να έχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα σε αυτές τις τόσο σημαντικές πολιτικές τη Ένωση, θα πρέπει να πιέσουμε και γειτονικέ χώρες ε, ε, ε, που εμφανίζουν ένταση και κινητικότητα επιθετική να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση πολύ περισσότερο δε εκείνοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή οικογένειά μας. ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, οι υπόπτες διασποράς απειλούν κυρίως τους αμάχους γιατί χρησιμοποιούνται σε περιοχές που δεν είναι ορατές. Ήδη υπόθηκε ότι το 78% των θυμάτων είναι άμαχοι και το 27% από αυτούς είναι παιδιά. Το μεγαλύτερο μέρος από τις βόμβες διασποράς δεν εκρήγνεται κατά την πρόσκρουση και παραμένουν στο έδαφος. Πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παρόλα αυτά δεν υπέγραψαν τη σύμβαση για τις βόμβες διασποράς γιατί έχουν τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα. Πράγμα ε, ιδιαίτερα ε, λυπηρό. Συμφέροντα που έχουν σχέση με την παραγωγή και την πώληση αυτών των όπλων. Δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση πιστεύω ότι τα ανθρωπιστικά συμφέροντα και η προστασία των αμάχων θα πρέπει να παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να επιμείνει έτσι ώστε όλα τα μέλη να υπογράψουν τη σύμβαση για τις βόμβες διασποράς. Ευχαριστώ τον κύριο Νικολάτσικ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κέλλη. Μιλήσαμε για την φεά πλευρά της σύγχρονης ζωής. Την ανθρώπινη καταστροφή από το HIV-AIDS. Τώρα μιλάμε για την καταστροφή των αθών πολιτών από τα πυρομαχικά διασπόρας. Ας προσπαθήσει η Βαρόνια από τη θέση της να δώσει κάποιες λύσεις. Αλλά το πρόβλημα βέβαια είναι να φτιάξουμε και τα πράγματα στην Ευρώπη. Μόνο 11 χώρες να έχουν υπογράψει δεν είναι σωστό. Πρέπει λοιπόν να πιέσετε έτσι ώστε να ζητήσετε από τις υπόλοιπες χώρες να απομακρύνουν τα εμπόδια που υπάρχουν για την επικύρωση της συνθήκης. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ομιλεί με μία φωνή στον υπόλοιπο κόσμο. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, αν δεν φτιάξουμε τη δική μας αυλή, πώς μπορούμε να δίνουμε μαθήματα στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μπορούμε να παίξουμε ε, τον ρόλο του σωστού παραδείγματος. Επαναλαμβάνω λοιπόν, να διορθώσουμε τα δικά μας προβλήματα πρώτα και μετά να ασχοληθούμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Τι θα κάνετε έτσι ώστε οι 16 χώρες να επικυρώσουν πριν από την 1η Αυγούστου. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Έχω σημειώσει τις ανησυχίες σας και τις παρατηρήσεις σας. Ξεκινώντας θα πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να επιμένει στην πλήρη κατάργηση και απαγόρευση των πυρομαχικών αυτού του τύπου μέσω των συμβάσεων για τα συμβατικά όπλα, των συνθήκων για τα συμβατικά όπλα. Θα συνεχίσουμε επίσης ε, να οργανώνουμε τη δράση μας ε, εναντίον αυτού του τύπου των πυρομαχικών στα πλαίσια της πολιτικής βοήθειας για την ανάπτυξη. Πρώτον, η, η απόφαση για την ένταξη στην συνθήκη αυτή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο φυσικά θα πρέπει να υποστηριχθεί και από τα κράτη-μέλη, είναι δική τους αρμοδιότητα και είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουν όλοι προσεκτικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε αυτή τη στιγμή 11 χώρες που έχουν υπογράψει και επικυρώσει, αλλά έχουμε άλλες 8 οι οποίες έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν ακόμα επικυρώσει. Συνολικά έχουμε 19 χώρες λοιπόν που έχουν υπογράψει. Και έχουμε και 8 χώρες που δεν έχουν κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τα μέλη λοιπόν ξεκαθάρισαν ότι θέλουν ε, τον μέγιστο δυνατό αριθμό χωρών να προχωρήσουν στην υπογραφή και επικύρωση. Θα ήθελα επίσης σύντομα να σταθώ σε αυτό που είπε η κυρία Λίν για τη βοήθεια στις τρίτες χώρες. Όπως είπα στις προηγούμενες παρατηρήσεις μου, θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις τρίτες χώρες στα πλαίσια της πολιτικής μας και της αναδιοργάνωσής της, έτσι ώστε να τις καταστήσουμε πιο αποτελεσματικές. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και μέσω των πολιτικών μας εξωτερικής δράσης να συνεχίσουμε την προσπάθεια για τη διάθεση και εξουδετέρωση όλων αυτών των όπλων, είτε είναι εγκαταλελειμμένα είτε άχρηστα πλέον. Το είπε και η κυρία Λούνατσεκ, τι συμβαίνει όταν αυτά τα σφαιρίδια, τα πολύχρωμα εμφανίζονται στην επιφάνεια του εδάφου και υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά τα οποία έχουν ακροτηριαστεί, έχουν χάσει και τη ζωή τους. Θα χρησιμοποιήσουμε τα λεγόμενα γεωγραφικά μέσα τα οποία έχουμε, τις περιφερειακές πολιτικές, όπως επίσης και τα μέσα για ανθρωπιστική βοήθεια, όπως το κάνουμε στο Σρι στο Λίβανο, στην Καμπότζη κτλ. Αναφέρθηκα στο ότι ξοδεύουμε 332 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση, έχουμε δαπανίσει μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και στο Αφγανιστάν και στο Λίβανο. Έχουμε προγράμματα για τη Βοσνία, Ευζεγοβίνη, το Λάος και την Καμπότζη. Έδωσα κάποιους αριθμούς, αλλά είναι δύσκολο να ποσοστικοποιήσει κανείς τα προγράμματα αυτά γιατί ε, όταν ε, δραστηριοποιούμεθα επιτόπου δεν διαφοροποιείται το αποτέλεσμα από την συνολική προσπάθεια πολλές φορές. Θα ήθελα επίσης να πω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την ε, εύθετη χρονικά επικύρωση της συνθήκης αυτής, της σύμβασης αυτής από τα κράτη-μέλη τίθεται εδώ ένα θέμα καθολικότητας ε, της συγκεκριμένης αυτής σύμβασης. Αποφασίσαμε να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε περισσότερο και στην ε, Διευθυντική Επιτροπή η οποία θα συνέλθει το Σεπτέμβριο στη Γενέβη έτσι ώστε όταν έχουμε την πρώτη συνάντηση των εμπλεκομένων να υπάρξουν ήδη αποτελέσματα. Είναι μεν αργά, αλλά η συζήτηση είχε πολύ μεγάλη σημασία για όλους και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Άστον, έτσι έκλεισε η μας συνεδρίαση. Καλό βράδυ σε όλους.